Good evening to everybody. Καλησπέρα σας. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτή την διακοινοβουλευτική συνάντηση. Καλώς ορίσατε. Θα χωρίσουμε την συνάντηση σε δύο σκέλη. Το πρώτο που αφορά ε, την ε, ε, ισότητα στην Ευρώπη και το δεύτερο τους δίκαιους κατώτατους μισθούς. Πριν μπούμε στην ουσία θέλω να μιλήσω λίγο για τα οργανωτικά. Οι κάρτες για να ζητήσετε το λόγο υπάρχουν στην αίθουσα και όσοι εθνικοί οι ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε λευκές κάρτες που έχουν αυτή τη μορφή. Προσοχή όμως γιατί είναι ειδικέ. Άλλες είναι για, την πρώτο, για το πρώτο σκέλος και άλλες για το δεύτερο. Ε, ο χρόνος ομιλίας θα κατανεμηθεί ω εξή. Τρεις εθνικοί βουλευτές, θα ακολουθήσει ένας ευρωβουλευτή και κατόπιν άλλοι τρει ε, εθνικοί βουλευτέ κλπ. Βεβαίω, αυτό μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί στη διάρκεια της συζήτηση. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Κόρτον Μάρας που είναι ο επικεφαλής της ε, Επιτροπής Εργασίας, Συστήματος Ταξιοδότησης και Κοινωνικής Εταιρικής Σχέσης του, ε, του Κοινοβουλίου της Κροατίας για να κάνει την εισαγωγή του και θα αναλάβει την Προεδρία. Γεια σας, θα συνεχίσω να μιλάω, αλλά σουηδικά, παρακαλώ, ε, σου, ε, με συγχωρείτε, κροατικά, παρακαλώ να φορέσετε τα ακουστικά σας. Αγαπητή κυρία Νικολσόνοβα, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η ευκαιρία να απευθυνθώ σε ευρωβουλευτές και βουλευτές. Σας ε, καλωσορίζω όλους. Ως πρόεδρος αυτής της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσουμε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το ένα είναι η καταπολέμηση της φτώχειας με το οποίο και θα ξεκινήσουμε γιατί όλοι γνωρίζουμε τη σημασία της δημογραφικής εξέλιξης των προσπαθειών που καταβάλουμε να δημιουργήσουμε αν όχι ταυτόσιμα πρότυπα, τουλάχιστον παρόμοια πρότυπα για όλους τους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό, κυρίως ε, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού. Πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον όλοι. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε απαιτούν να κινηθούμε γρήγορα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνώρισε τη σημασία του ζητήματος. Υπάρχει κάποιος πλέον που έχει την άμεση ευθύνη της των δημογραφικών θεμάτων. Γι' αυτό το λόγο θα ε, περάσω τώρα το λόγο στην Επεύθυνη Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Μάρας. Αγαπητέ συνάδελφε κύριε Σμιτ, ε, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω εδώ και να κάνουμε και ανταλλαγή απόψεων για την εγγύηση τέκνου. Οι συνάδελφοι Τζεντιλόνι και Ντομπρόφσκης μίλησαν για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σήμερα το απόγευμα μαζί σα. Και σήμερα ε, ε, μιλήσαμε και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο το επόμενο εξάμεινο. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είπε ότι πρέπει ε, να μιλήσουμε περισσότερο για το μέλλον. Είναι σαφές αυτό. Δείχνει τη σημασία που αποδίδει η κυρία Φοντερ Λάιεν στα παιδιά και στην παιδική φτώχεια. Μαζί με τον Νίκολα Σμιτ, τον συνάδελφό μου, ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε την εγγύηση για αυτή για τα παιδιά το 2021 τα αξιότιμα μέλη παρόντα εδώ σήμερα θα συμφωνήσουν μαζί μου όταν πω ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην υποστήριξη που χρειάζονται κατά την παιδική του ηλικία και την εφηβεία. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών ε, βρίσκονται στο άρθρο 3 Τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Θέλω να υποστηρίξω και να συμπληρώσω τα κράτη-μέλη στο έργο τους για τα παιδιά. Το Νοέμβριο του 2017 το Κοινοβούλιο αυτό μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφάλισαν ότι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Αξιότιμα μέλη, κατά την ακρόασή μου πριν από λίγους μήνες, σε αυτό το κοινοβούλιο, όχι σε αυτή την αίθουσα όμως, δήλωσε ότι η προτεραιότητά μου ήταν να επενδύσω στα παιδιά. Ε, μένω προσκολλημένη στο στόχο μου και δηλώνω ότι χρειάζομαι την υποστήριξή σας για να ε, συμβούν όλα αυτά το 2013 είχαν γίνει συστάσεις σε σχέση με τη, τα μέτρα για τα παιδιά για να σπάσουμε τον κύκλο της μειονεξίας. Πρέπει να έχουμε γι' αυτό πρόσβαση σε κατάλληλους πόρους, σε αποτελεσματικές υπηρεσίες και να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των παιδιών να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστιθέμενη αξία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πάρει τη μορφή η ειδική εγγύηση τέκνων για την αντιμετώπιση των φυσταμένων φραγμών σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα αυτοί οι φραγμοί που εμποδίζουν τα παιδιά από την πρόσβαση σε υπηρεσίες που χρειάζονται για την καλή τους υγεία και την προσωπική τους ανέλυξη. Ε, Μία ολοκληρωμένη εγγύηση τέκνου θα ε, βοηθάει τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, θα διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ε, στέγης και βεβαίως ε, καλής διατροφής. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή αξιολογεί την ουσία της πρωτοβουλίας αυτής για την εγγύηση τέκνου. Σε λίγη ώρα ο συνάδελφος Νίκολα Σμιτ θα δώσει περισσότερα ε, στοιχεία για τους στόχους μας ε, σε αυτό τον κρίσιμο φάκελο. Επίσης, ε, ανέλαβα να ετοιμάσω μια συνεκτική στρατηγική για τα δικαιώματα των παιδιών. Είναι ακόμα νωρί σε αυτή τη διαδικασία, αλλά ο στόχος μας είναι να συμπεριλάβουμε δράσεις για να προστατεύσουμε τα ευάλωτα παιδιά online και offline, να ενισχύσουμε τη δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά και να προλάβουμε και να καταπολεμήσουμε τη βία. Θα χαρείτε, είμαι βέβαιη, να ακούσετε ότι αυτή η στρατηγική προωθεί και τη συμμετοχή των παιδιών στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Π.χ. υπό την αιγίδα, η ιδέα είναι υπό την αιγίδα για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης να συμπεριλάβουμε διάλογο, διαλόγους παιδιών και θερινές κατασκηνώσεις ε, με ορισμένα θέματα που θα προτείνονται από τα παιδιά. Η Κομισιόν ε, προχωράει στο, με το πρόγραμμα πίσω στα σχολεία. Θέλουμε να αυξήσουμε επίσης την προστασία των μεταναστών παιδιών και των ασυνόδευτων ε, ανήλικων. Είναι από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους αυτοί στην κοινωνία μας σήμερα, αγαπητά μέλη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραλείψουμε μια γενιά παιδιών. Έχουμε ισχυρή θεσμι... Ε, νομική βάση, το άρθρο 3.3 για παράδειγμα της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 24 και 32 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τα Δικαιώματα του Παιδιού το από το 2011 ε, εξακολουθεί να ισχύει, όπως και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν προσυπογράψει. Ε, βεβαίως χρειάζεται ευρία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους ε, την κοινωνία των πολιτών, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να δούμε τι κάνουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε για τα παιδιά μας. Θέλω επίσης να ακούσω από τα ίδια τα παιδιά, όπως είπα, τις απόψεις τους, τις ανάγκες τους. Πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Η στρατηγική θα εγκριθεί μάλλον στο πρώτο εξάμεινο του 2021. Και αγαπητά μέλη, κάποτε υπήρξαμε όλοι παιδιά. Είναι ζωτική σημασία κάθε παιδί να έχει δικαίωμα και πρόσβαση σε ε, ε, ισότιμες συνθήκες κατά την αρχή της ζωής του. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή τους στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Αξιότιμα μέλη, το έργο μας στηρίζεται στο Μηχανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ευθυγραμμιζόμαστε με την ατζέντα του 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη του ΙΕ. Η στρατηγική έχει τη δυνατότητα να ε, προσδώσει προστιθέμενη αξία στα, στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, γιατί θα έχουμε ένα ε, ισχυρό αφήγημα που θα λάβουμε υπόψη μας στις συζητήσεις μας στα πολυεθνικά φόρα. Πάντοτε να θυμόμαστε ότι τα δικαιώματα των παιδιών είναι καθολικά και το παιδί παραμένει παιδί ανεξάρτητα από το που βρίσκεται και μεγαλώνει σε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Σουίτσα. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, εισαγωγική σας ε, αυτή τοποθέτηση και ελπίζω το σχέδιο να προβλέπει και πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο και την επιγραμμική τους προστασία. με πήρε τηλέφωνο το προηγουμένω η κόρη μου και δεν μου είπε μπαμπά σ' αγαπώ, είπε μπαμπά έχει πέσει το διαδίκτυο. Και ε, τώρα ε, ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Νικολά Σμιτ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Ας αρχίσω με ε, το εξή. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να συμμετέχω στη συζήτηση αυτή για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αξιότιμα μέλη, γεννήθηκε η ίδια ιδέα της εγγύηση για τα παιδιά. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ε, ότι συμμετείχα το 2015 σε σεμινάριο όπου προείδρευε ένας από τους συναδέλφους μας εδώ ως εκπρόσωπος της τότε Προεδρίας του Λουξεμβούργου όταν κατατέθηκε αυτή η ιδέα. Και όπως γνωρίζετε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είπε και η συνάδελφός μου, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ε, υποσχέθηκε να οικοδομήσει σε μια νέα ιδέα για την εγγύηση για τα παιδιά και να υποστηρίξει κάθε παιδί ε, που έχει ανάγκη έχω την τιμή να είμαι αρμόδιος για την εκπόνηση αυτού του έργου μαζί με το πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και το πρόγραμμα δράσης του. Θα συνεργαστώ στενά με την Αντιπρόεδρο Σουίτσα, η οποία ε, έχει την ηγεσία σε αυτά τα θέματα της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και θα καταθέσουμε μια συνολική στρατηγική, όπως σας είπε, για τα δικαιώματα των παιδιών. Τα, η παιδική φτώχεια είναι άδικη αρχή για τη ζωή ενός παιδιού. Η φτώχεια όμως ε, επηρεάζει τους πάντες σε μια φτωχή οικογένεια και τους γονείς και τα παιδιά. Τα φτωχά παιδιά συνήθως ζουν σε φτωχές οικογένειες. Και ε, γι' αυτό θέλουμε να δούμε και τη δράση μας για τα φτωχά παιδιά ε, να εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης της φτώχειας. Αν καταπολεμήσουμε τη φτώχεια των γονέων, βελτιώσουμε τη ζωή τους και τους δώσουμε τις κατάλληλε ευκαιρίες, τότε υποφελούνται και τα παιδιά. Επόμενο. Άρα χρειάζονται και οι γονείς καλές δουλειές, αξιοπρεπείς, ίσες ευκαιρίες για όλους, ε, με ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να βρουν καλύτερη δουλειά χρειάζονται και συνθήκες εργασίες δίκαιες. Θα συζητήσουμε στην επόμενη ενότητα το δίκαιο κατώτατο μισθό. Επιτρέψτε μου να σας πω από τώρα ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που βοηθάει να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή γονείς και παιδιά. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σωστή κατάλληλη κοινωνική προστασία και πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα επίσης σημαντικό εργαλείο πολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού. Ε, η αρχή 11 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων ήταν επίσης έμπνευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δική σας δηλαδή, και ε, φωτίζει τα δικαιώματα των παιδιών σε ποιοτική μόρφωση και σε καλή ε, προσχολική ηλικία. Επίσης αναφέρεται το δικαίωμα των παιδιών να προστατεύονται από τη φτώχεια, από τον κίνδυνο της φτώχειας. Παιδιά που είναι από μειονεκτικές ε, συνθήκες, οι μειονεκτούσες οικογένειες θα πρέπει να έχουν τις ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες. Εκεί η εγγύηση για τα παιδιά μπορεί πραγματικά να προσθέσει ε, ουσιαστική υπεραξία. Είναι πολύ ψηλός σήμερα ο αριθμό των παιδιών που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2018 περίπου 19 εκατομμύρια παιδιά ζούσαν στη φτώχεια στα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης. Ήδη, ε, ε, τότε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλο, Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και αυτό πρέπει να προσθέσετε άλλα 4 εκατομμύρια, 23 συνολικά. Η παιδική φτώχεια μπορεί να είναι πιο υψηλή σε κάποια κράτη-μέλη σε σχέση με άλλα. Υπάρχει όμω ένα κοινό χαρακτηριστικό. Σε όλα τα κράτη-μέλη παρατηρείται, ακόμα και στα πλούσια κράτη. Γι' αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε ένα εργαλείο πολιτικής που να πυροδοτήσει δράσεις από τα κράτη-μέλη τι προτεραιότητε των πολιτικών και την εξασφάλιση επαρκούς εθνικής χρηματοδότησης. Η Ένωση μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια αυτή με καινοτόμε προσεγγίσεις, με υποστήριξη των σωστών επενδύσεων και ε, υιοθετώντα αυτό το καινοτόμο κατάλληλο πλαίσιο μαζί με τα κράτη-μέλη και έτσι να σφυριλατήσει τη δράση και τα θετικά μέτρα επί τόπου έτσι ώστε να είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Προετοιμάζοντα λοιπόν ένα τέτοιο εργαλείο πολιτικής, συμμερίζομαι απολύτω τη δική σας δέσμευση. Θα πρέπει να εστιάσουμε στα παιδιά που έχουν ανάγκη και στην πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. Ε, θα πρέπει να επενδύσουμε, ας πούμε, σε ποιοτική εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία, ε, φροντίδα στα σχολεία, ε, πρόσβαση στην υγεία, στη διατροφή και σε αξιοπρεπή στέγη για να σπάσει ο φαύλος κύκλος ε, της μειονεξίας που αντιμετωπίζουν τα φτωχά παιδιά. Θα πρέπει με προσοχή να κάνουμε το καθήκον μας για να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό μέσον. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα βασιστεί στις μελέτες αντικτύπου που ζήτησε το Κοινοβούλιο και σκοπιμότητας. Η πρώτη μελέτη κατατέθηκε τη Δευτέρα και θα μας βοηθήσει να ε, ορίσουμε και να σχεδιάσουμε τις σωστές πολιτικές. Η εγγύηση για τα παιδιά θα είναι ένα από τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τον αποκλεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σας είπα προηγουμένως, όταν τα μέτρα είναι προ όφελο των γονέων, είναι και προ όφελο των παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσης θα έχει μια προσέγγιση συνολική κατά της φτώχεια, υποστηρίζοντας τα κράτη-μέλη που πατάσουν τη φτώχεια. Η εγγύηση λοιπόν για τα παιδιά θα είναι ένα βασικό κεντρικό ε, στοιχείο, μια ψηφίδα αυτού του ε, του Ευρωπαϊκός πυλώνα ε, Κοινωνικών Δικαιωμάτων και εφαρμογή του, Επίση, πολύ σημαντικό και οι διάφορες αρχές του μα εμπνέουν για να σχεδιάσουμε πολιτικέ κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, υπέρ τη αξιοπρεπούς εργασία, των θέσεων εργασία, επενδύσεις, κοινωνική προστασία, ε, κοινωνικές υπηρεσίες, προσιτές και κυρίως προσιτή κατοικία. Το 2021 θα καταθέσουμε την εγγύηση για τα παιδιά μετά τις απαραίτητες ε, προεργασίες και μεταξύ αυτών θα είναι και η διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και ενεχομένους και θα επωφεληθούμε και από τις προπαρασκευαστικές δράσεις και την τρέχουσα διαβούλευση για μια ε, ισχυρή Ευρώπη στη δίκαιη μετάβαση. Η προπαρασκευαστική δράση που έχει προτείνει το Κοινοβούλιο και τώρα εκτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο έργο μας. Θα συνεχίσουμε επίσης το, τα πολύτιμα πιλωτικά ε, προγράμματα και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Τρέχουν ακόμα. Εχθές ήμουν σε μια διάσκεψη που έκλεισε την πρώτη φάση των προπαρασκευαστικών δράσεων και κατέθεσε την πρώτη μελέτη σκοπιμότητας. Η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση θα ακολουθήσουν. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα στήριξης ε, χρηματοδοτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Αξιότιμοι βουλευτές, πέρσι τον Απρίλιο σε ένα ψήφισμά σας τονίσατε ότι η εστίαση στη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, ΣΥΝ θα πρέπει να αφορά τα πιο φτωχά παιδιά με έμφαση στις υπηρεσίες. Ζητήσατε 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το έκτηση να ε, αφιερωθούν στην εγγύηση ε, για τα παιδιά. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, να δίνουν τουλάχιστον το 5% των πόρων τους από το ΕΚΤΣΙΝ για να υλοποιήσουν τις συστάσεις του 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επένδυση στα παιδιά. Θα παρακολουθώ πάρα πολύ στενά τους τριμερείς διαλόγους για αυτά τα θέματα, αλλά δεν ξεκινούμε από μηδενική βάση. Τα ευρωπαϊκά ταμεία ε, κονδύλια ήδη βοηθούν πάρα πολλά παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Στόχος μας είναι να βρούμε τους απαραίτητους πόρους για να υποστηρίζουμε τα παιδιά αυτά που το έχουν ανάγκη. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από μόνη της δεν θα είναι αρκετή για να βγουν τα παιδιά, τα εκατομμύρια των παιδιών από τη φτώχεια. Χρειάζεται και εθνική ενίσχυση. Θα πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί αυτή η εγγύηση για ε, τα παιδιά ε, και έχουν το ρόλο τους και τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία σήμερα εκπροσωπούνται εδώ. Είναι πρωταγωνιστικός αυτός ο ρόλος. Αν είναι καλά στοχευμένα όλα και αν υπάρχουν και οι δυνατότητες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Invest EU θα εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνέργειες και θα κάνουμε την αλλαγή. Πάνω από όλα όμως χρειαζόμαστε μια ισχυρή δέσμευση σε όλα τα επίπεδα, κοινή, ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό, να επενδύσουμε στα παιδιά μας για μια δίκαιη κοινωνία βιώσιμη και ανθεκτική. Μία από τις προτεραιότητες μας είναι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, όπως είπε η Αντιπρόεδρος Σουίτσα, αλλά και η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό θα αναφέρεται και στις συστάσεις αναχώρα που θα εκδώσουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που προηγουμένως συζητήσατε. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα τα συζητούμε όχι μόνο με τις κυβερνήσεις αλλά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών και τις ε, αρχές της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή με όλους τους ενδιαφερομένους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Νικόλα Σμιτ, ε, Ευρωπαίο Επίτροπο θέσεων εργασίας και, κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντουάρτο Μπαρόκοντε Μέλο, μέλος του Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας. Αξιότιμη Συμπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Κορατική Προεδρία, αγαπητέ Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για θέματα δημοκρατία και δημογραφία, ε, αγαπητέ ε, Επίτροπε, Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές ε, που προσκάλεσαν την Πορτογαλία να συμμετάσχει σε αυτή τη συνεδρία. Η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ επίκαιρη και τι αποκαλύπτει πώς έχει μετακινηθεί η προσοχή από τα θέματα των δημοσίων οικονομικών και της λιτότητας των τελευταίων χρόνων προς ε, το θέμα της κοινωνικής Ευρώπης και της ε, δίκαιης μετάβασης. Είναι πάρα πολύ θετικό που υπάρχει αυτή η ιδέα για την εγγύηση για τα παιδιά και οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που σημαίνουν ότι η δράση δράσει μα βρίσκονται στην καρδιά όλων των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθε ε, οργάνωσε μια ε, διάσκεψη για το θέμα τη εγγύηση για το παιδιό και Πράγμα που σημαίνει ότι θα μας δώσει χρόνο ε, για το, να συζητήσουμε τα θέματα. Η, παιδική φτώχεια είναι κάτι το οποίο μετράται ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών ζουν σε, ε, σε φτώχεια, 8,5% συγκεκριμένα, 9,3% ε, ζουν σε οικογένειες χωρίς που δεν εργάζονται και το 2,5% ζουν και ε, στις τρεις αυτές προϋποθέσεις. Αυτό επηρεάζει όλα τα κράτη. Σας παρακαλούμε, λέει ο Πρόεδρος, να μιλάτε λίγο πιο αργά, να διαβάζετε λίγο πιο αργά υπάρχουν ε, μεγάλες διακυμάνσεις ε, από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Τα στοιχεία του 2014 δείχνουν ότι τα παιδιά της Ρουμανίας και στην Βουλγαρία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχει 20%. Σας παρακαλώ πιο αργά επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος. Η παιδική φτώχεια ως εκ τούτου είναι ένα πρόβλημα όλης Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πηγή ανισοτήτων το 2013 το ε, Συμβούλιο ενέκρινε την σύσταση επενδύοντας για τα παιδιά που έδωσε έμφαση στην απασχόληση. Το 2017 μόνο, μέχρι το 2017 μόνο εννέα κράτη-μέλη είχαν λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματα αυτά. Ως εκ τούτου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 2015 ε, ενέκρινε ένα ψήφισμα που ζητούσε την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά που επιβεβαιώθηκε πιο πρόσφατα με ένα ψήφισμα ε, για το ε, esf ε, ΣΥΝ που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2019. Στη χώρα μου έχουμε φτώχεια μεγαλύτερη στην ηλικίες 0 έως 18 από ό,τι οι άλλες ηλικίες. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την παιδική φτώχεια με την εξέλιξη και προσπα των πολιτικών μας. Επίσης θέλουμε να διευρύνουμε την γονική άδεια να επενδύσουμε σε καλύτερα προγράμματα στέγασης μεταξύ άλλων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πεπισμένοι ότι η εγγύηση για τα παιδιά θα πρέπει να είναι μια νέα προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές πλευρές της παιδικής φτώχειας. Γιατί κάθε παιδί ε, στην, που κινδυνεύει από φτώχεια θα, έχει, θα πρέπει να έχει ανάγκη σε ποιοτική εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, ε, σχολική ε, καλά σχολεία και ε, μια σειρά από άλλες ε, παροχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να συμφωνήσει για δεσμευτικούς δείκτες ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα που έχει πολλές διαστάσεις θα πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέλος κομμάτι του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα πρέπει να ε, περιληφθεί σε συγκριτικούς δείκτες ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν με βάση αυτούς να ε, ε, να διατυπώνουν ολοκληρωμένα προγράμματα. Η εγγύηση για τα παιδιά θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Υπάρχει ένας ένας, ε, ένα ποσό του προϋπολογισμού 5,9 δις και θα πρέπει αυτός να χρησιμοποιηθεί σωστά. Βεβαίως μας απασχολεί το γεγονός ότι στο πρόσφατο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει μειωθεί το ποστό κατά 1,7 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μικρότερο από την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική όθηση για την εγγύηση για τα παιδιά που προέκυψε από την πρόταση της κυρίας Φόντερ θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με, το, με τα ποσά του ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να, ε, να αναπτυχθούν προγράμματα παροχή υγειονομικής περίθαλψης, η εκπαίδευση και η στέγαση, ας πούμε. Για να, να επιτύχει το πρόγραμμα αυτό εγγύησης για τα παιδιά θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμμετάσχουν αποτελεσματικά η εγγύηση για τα παιδιά θα πρέπει να είναι βασικό μέσο για μια θετική αλλαγή στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και ευκαιρία της ε, παρουσίας της Αντιπροέδρου. Θα ήθελα να προτείνω όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε εδώ να επισέλθουν στο κέντρο της συζήτησης της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης που θα ξεκινήσει σε 9 Μαΐου. Αποτελεί μοναδική ευκαιρία ώστε οι νέοι Ευρωπαίοι που είναι και το μέλλον μας να έρθουν στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστώ. Προχωρούμε τώρα στους ομιλητές ε, που γνωρίζουν ότι διαθέτουν δύο λεπτά χρόνο. Ο κύριος Βόικος από τη Σλοβενία. <laughs> Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα σλοβενικά. Χαίρομαι πολύ που ακούω ότι μία προτεραιότητα για την Κομισιόν αυτή είναι ο κοινωνικός πυλώνας των δικαιωμάτων. Αυτό σίγουρα θα συμβάλλει σε μια δικαιότερη, πιο αλληλέγγυα Ευρώπη, πιο ολοκληρωμένη. Επίσης χαίρομαι πολύ που σας άκουσα να μιλάτε για την εγγύηση τέκνου ιδιαίτερα για τα παιδιά τα μειονεκτικά, από μειονεκτικές ομάδες. Τα μειονεκτήματα πλήττουν τα παιδιά σε όλα τα επίπεδα. Η φτώχεια επηρεάζει και τη σωματική και την ψυχική ανάπτυξη. Μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου, όπως απέδειξε η έρευνα στην ευρωψυχολογία. Δεν είναι μόνο έλλειψη υλικών αγαθών, Πρόκειται για έλλειψη κοινωνικού κεφαλαίου για των φτωχών παιδιών, αγοριών και κοριτσιών. Και σίγουρα δεν αρχίζουν τη ζωή τους επίσης ώρες. Η φτώχεια ε, επηρεάζει τα παιδιά που έχουν γεννηθεί φτωχά Αυτά τα παιδιά έχουν πρόβλημα σε όλη τη ζωή τους, γιατί δεν απολαμβάνουν τα προνόμια άλλων παιδιών. Στο σχολείο επίσης δεν είναι ισότιμα με τους ε, συμμαθητές. Πολλές φορές ε, υποφέρουν από κοινωνικό ε, αποκλεισμό και δεν αναπτύσσουν το δυναμικό τους. Περιορίζονται από τις ικανότητες, δυνατότητες της οικογένειας και δημιουργείται φαύλος κύκλος που δυσκολεύει τη ζωή. Για τη Σλοβενία χαίρομαι μπορώ να πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία ε, στοιχεία της Eurostat, ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για τα παιδιά στη Σλοβενία είναι, ο κίνδυνος είναι ο χαμηλότερος σε σχέση με όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Παρόλα αυτά είναι στο 13,1% που είναι υψηλό ποσοστό. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ αξιότιμε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πρωτίστως θέλω να πω πόσο χαίρομαι που μπορώ να συμμεριστώ τις απόψεις μου για αυτό το σημαντικό θέμα που αποτελεί τόσο σημαντικό καθήκον για τους Ευρωπαίους συνομοθέτες κατά αυτή τη θητεία. Η Βουλγαρία είναι υπέρ της ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπ' αυτή την έννοια ε, τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι τεράστια σημασίας η πρωτοβουλία για την ενίσχυ... Ε, ε, εγγύηση τέκνου είναι η κύρια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη... είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για τη Βουλγαρία όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι το κύριο κοινωνικό θέμα, ήταν επί Βουλγαρικής Προεδρίας το 2018 και δεχτήκαμε πολλά συμπεράσματα του Συμβουλίου για την μείωση της φτώχειας και την αύξηση της κοινωνικής ένταξης. Ε, ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση ε, χτίσαμε την πολιτική μας για τα παιδιά, τη φροντίδα των παιδιών που είναι από τις βασικές μεταρρυθμίσεις που κάνουμε στην Βουλγαρία και επίσης προσέχουμε και τις υπηρεσίες για την πρώιμη παιδική ηλικία με εστίαση στα παιδιά μέχρι 7 ετών, παιδιά με αναπηρίες και τις οικογένειές τους, όπως και τους ε, μελλοντικού γονείς. Πιστεύουμε ότι μόνο μια οριζόντια σύνθετη προσέγγιση που γίνεται σε εταιρική σχέση με άλλους εμπλεκομένους μπορεί να δώσει θετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό η Βουλγαρία είναι έτοιμη να συμμετάσχει ενεργά και να συμβάλλει στη διαδικασία των νέων πρωτοβουλειών για την εγγύηση τέκνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο Στην κυρία Βίτα Γκρόσα Ζαλίτα από τη Λετωνία. Can you, can you open uh, uh the mic? Yeah. Thank you. Ευχαριστώ. Ε, μιλώ εξ ονόματος της Λετωνίας. Τα τελευταία χρόνια συγκέντρωσε πολύ μεγάλη ε, προσοχή ε, και εστίασε την προσοχή της ιδιαίτερα ε, για οικογένειες που έχουν πρόβλημα. Πάντα αυτές θα είναι προτεραιότητα στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις οικογένειες αυτές. Όταν μιλούμε για εγγυήσει, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε όλη την Ευρώπη να υπάρχουν αντίστοιχες δυνατότητες παντού σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην υγεία, ε, στη στέγη, ε, ε, στην εκπαίδευση, στα σχολεία. Εδώ χωράει πολλή δουλειά. Πολύ συχνά η φτώχεια κληρονομείται από τη μια γενιά στην άλλη. Και αυτά είναι μεγάλα προβλήματα και κίνδυνοι που πρέπει να μας απασχολήσουν. Η εγγύηση για τα παιδιά θα πρέπει να ειδωθεί σε ευρύτερο επίπεδο, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό. Όσο πιο ισχυρές είναι οι οικογένειες, τόσο ισχυρότερη θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Λετωνία εργαζόμαστε έτσι ώστε κάθε παιδί να μπορεί να μεγαλώνει μέσα στην οικογένειά του. Έχουμε διάφορα ε, σχέδια αλλά είναι πολλά τα προγράμματα και πολλά τα προβλήματα. Φυσικά και η λύση θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία ε, Μπλίνκεβιτσούτε, αντιπρόεδρο Επιτροπή ε, Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση να σας κάνω πρώτα απ' όλα. Χρειάζεστε πραγματικά μια ευρωπαϊκή εγγύηση για την νεολαία. Όποιον και να ρωτήσετε, επιτρόπους, μέλη εθνικών κοινοβουλίων, θα σας απαντήσουν ότι βεβαίως και χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή εγγύηση για την νεολαία και είναι υψή τη σημασία. Φαίνεται τόσο στοιχειώδες, τόσο ευνόητο, τόσο αυτονόητο. Κάθε παιδί, όπου και αν ζει στη Λιθουανία, ε, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Κροατία, στη Σλοβενία. Κάθε μικρό παιδί έχει το δικαίωμα ε, σε ποιοτική εκπαίδευση, σε υπηρεσίες υγείας, σε στέγη, σε σωστή διατροφή. Όλα αυτά είναι στοιχειώδη. Όμως αγαπητοί μου φίλοι, εμείς είμαστε πολιτικοί. Γιατί είναι περίπου 20 εκατομμύρια τα φτωχά παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια ε, κοινότητα που είναι πάρα πολύ πλούσια και δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχειώδη που σας ανέφερα. Ο Νίκολα Σμιτ είπε ότι πριν από πέντε χρόνια ξεκινήσαμε αυτή τη σταυροφορία και επαναλαμβάνουμε έκτοτε ότι χρειάζεται αυτή η παιδική η εγγύηση για τα παιδιά. Θυμάμαι στην περασμένη θητεία ότι πιέζαμε διάφορες πολιτικές ομάδες ακριβώς για να πετύχουμε να μας υποστηρίξουν και άλλες πολιτικές ομάδες, τα δικά μας ψηφίσματα. Δεν αρκεί να έχουμε εθνικά ταμεία, εθνική χρηματοδότηση, εθνικές προτάσεις. Αυτό θα πρέπει να το ξεπεράσουμε και να φτάσουμε ε, σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μόνο έτσι θα καταπολεμηθεί η παιδική φτώχεια. Θυμάστε τη στρατηγική 2020 Υποτίθεται ότι θα είχε εκμηδενιστεί η φτώχεια μέχρι το 2020. Μόνο ένα εκατομμύριο παιδιά καταφέραμε να βγάλουμε από τη φτώχεια. Θα πρέπει να συνεργαστούμε, είναι προφανές αυτό. Και θέλω να πω προς τους εθνικούς βουλευτές ότι αυτό τον καιρό συζητούμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και αν παραμείνει η ελλειπής χρηματοδότηση που υπάρχει σήμερα, είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά θα συνεχίσουν να ζουν μέσα στη φτώχεια και δεν πρόκειται να δημιουργηθεί ποτέ η κοινωνική Ευρώπη. Σας ζητώ την υποστήριξή σας και τη συνεργασία σας για να σώσουμε τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Thank you very much for this emotional... Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ε, συγκινητική παρέμβαση. Μ' αρέσουν οι συναισθηματικοί πολιτικοί. Είναι πολύ καλό πράγμα αυτό. Ο κύριος Άντεμ Μπάβιτς από την Κροατία. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση ε, για το σημαντικό αυτό θέμα που αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντιμετωπίσει γύρανση του πληθυσμού και αρνητική φυσική εξέλιξη και χαίρομαι πολύ που υπάρχει αντιπρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέματα δημογραφία και δημοκρατία. Τα θέματα της, ε, αυτά ρυθμίστηκαν ε, νομικά στην Κροατία. Υπάρχουν τα δικαιώματα του παιδιού για την περίοδο 14-20 και έτσι έχουμε μεγαλύτερη προστασία της πρόθεσης και προστασίας του παιδιού ο στόχος της στρατηγικής που εκπονήθηκε είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεργαστούν για την ε, εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, για να, για εντοπίσουν ε, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και να καθορίσουν τις εθνικές προτεραιότητες και τους στόχους, ξεκινώντας με τη, από τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του παιδιού του 2015 η Ευρωπαϊκή, το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των παιδιών η στρατηγική αυτή έχει σκοπό την πλήρη επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Ε, ε, φιλικές προς τα παιδιά πολιτικές σε πέντε τομείς. Δικαιοσύνη, υγεία, ε, κοινωνική επιδική ε, πολιτική, παιδεία και αθλητισμός. Επίσης, κάθε, εξάλληψη κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών. Τρίτον, εξασφάλιση των παιδιών σε ευάλωτες καταστάσεις και τέταρτον, ίση συμμετοχή των παιδιών. Όπως είπε και ο κύριος Σμιτ στην εισαγωγική του ομιλία, θα, θα υπογραμμίσω και εγώ ότι η την εγγύηση των δικαιωμάτων των παιδιών με ειδικέ ανάγκες ε, σε παιδεία, στην αποκατάσταση, στην κοινωνική φροντίδα, σε εξατομικευμένο περιβάλλον όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη. Τα θέματα των... Ε, αυτά της αναπηρίας είναι πολύ ε, σημαντικά. Υπάρχουν τοπικές κοινότητες που έχουν διαφορετικά οικονομικά μέσα. Πρέπει λοιπόν να πω ότι συνολικά η πρόοδος είναι θετική, αλλά πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ιδίως στην προστασία των παιδιών σε ιδρύματα, παιδιών με αναπηρία και παιδιά που ζουν με φτωχές οικογένειες. Πιστεύω ότι ο επόμενος προϋπολογισμός θα μπορέσει να ε, χρηματοδοτήσει ε, δραστηριότητες που σχετίζονται με την εγγύηση για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Ε, η επόμενη ομιλήτρια η κυρία Σκέβη Κούτρα Κουκουμά από την Κύπρο. Σας ευχαριστώ. Η πρόταση για καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά αποτελεί μονόδρομο απέναντι στα δεδομένα που δείχνουν ότι ένα στα τέσσερα παιδιά βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν πρόκειται όμως απλά για ένα μεγάλο αριθμό. Πρόκειται για έναν έγκλημα απέναντι στη νέα γενιά και το μέλλον της Ευρώπης 25 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 ετών στερούνται ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την παιδική μέρημνα, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, υποσυτίζονται, είναι άστεγα ή στεγάζονται σε κακές συνθήκες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υποκρισία από πλευρά της Ευρώπης. Η παιδική φτώχεια δεν γεννήθηκε σε μια νύχτα και δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικών ξένων προ τι κατευθυντήριε γραμμέ τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί σήμερα όλοι και όλες να σημειώνουμε την ανάγκη για να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τη φτώχεια, αλλά δεν ήμασταν όλοι στο ίδιο στρατόπεδο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν επιβάλλονταν μια σειρά από μέτρα λιτότητα, τα οποία μείωναν του μισθού και το ονόμαζαν ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα, όταν προτείνονταν οριζόντιε περικοπέ στι κοινωνικέ παροχέ, γνωρίζοντα ότι αυτό θα άφηνε εκτεθειμένε και αβοήθητε δεκάδε χιλιάδε οικογένειε, όταν τερματίζονταν τα στεγαστικά προγράμματα για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να φτάσουν του οικονομικού στόχου των μνημονίων, όταν προγράμματα στήριξη μαθητών με αναπηρία ή μεταναστευτικό βιογραφικό είχαν περίπου εκλείψει από τη δημόσια παιδεία. Η αύξηση της παιδικής φτώχειας υποθηκεύει το μέλλον του κόσμου ολόκληρου. Τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχουν λιγότερες πιθανότητες συγκριτικά με τους πιο ευκατάστατου συνομιλίκους του, να έχουν καλή επίδοση στο σχολείο, να είναι υγιεί και να αναπτύξουν πλήρω τι δεξιότητε και δυνατότητε του ω ενήλικε. Δεν χρειάζονται συνέδρια και διασκέψει. Πολιτική βούληση χρειάζεται που η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώ δεν έχει λόγω ιδεολογικού προσανατολισμού. Που δυστυχώ μέσα από μεγαλόστομε διακηρύξει προσπαθούν να δείξουν ότι νοιάζονται. Που εξαγγέλνει κονδύλια που χάνονται στι διαδρόμου τη γραφειοκρατία και δεν φτάνουν στα παιδιά Ας σταματήσουμε να στρουθοκαμιλίζουμε και να πάρουμε αποφάσεις για έργα. Ευχαριστώ. Thank you very much. The next one is... Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άχνες Χονκέριος από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Thank you. Uh, thank you for uh, show. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας ήρθατε γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να συζητούμε για αυτά τα θέματα για την πρόληψη της παιδικής φτώχειας και να μην συζητούμε απλώς για το τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στα διάφορα επίπεδα και σε εθνικό επίπεδο και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Θέλω να τονίσω κάτι που είπε ο Επίτροπος Σμιτ, ότι η παιδική φτώχεια δεν αφορά μόνο τα φτωχά κράτη-μέλη, αλλά παρατηρείται και σε πλούσια κράτη-μέλη. Εγώ είμαι από τις κάτω χώρες. Έχουμε και στην Ολλανδία φτωχά παιδιά και αυτό πραγματικά είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Ακούσαμε και τους αριθμούς. Και όταν ξεκινάς τη ζωή σου στη φτώχεια, έχεις ένα μειονέκτημα από χέρι για όλη τη ζωή σου. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να πιέσουμε. Πώς να το πω τώρα. Όσους συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση που θα γίνει ε, τούτη εδώ την Πέμπτη στο Συμβούλιο που θα ασχοληθούν με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και πάλι ντρέπομαι ως Ολλανδή γιατί ένας από τους πρωθυπουργούς που τα έχει στυλώσει είναι ο δικός μας. Μόνο τον προϋπολογισμό κοιτάει και θέλει 1% ε, του ΑΕΠ μόνο να δίνεται στον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αντί να κοιτάει τις ανάγκες ε, και πώς αυτές θα καλυφθούν. Πώς μπορούμε εμείς να ενισχύσουμε την έκκλησή μας για την εγγύηση για τα παιδιά και εμείς στο ευρωπαϊκό επίπεδο ε, έχουμε ήδη ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά πώς θα συνεργαστούμε με το εθνικό επίπεδο για να υποστηρίξουμε τη ζωή των μικρών παιδιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρώσα Εστάρας από το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους και φυσικά και τους προέδρους. Λοιπόν, είναι σαφές ότι το θέμα των ανηλίκων και των παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα τα παιδιά που έχουν ε, αναπηρίες και ειδικέ ανάγκες. Αν θέλουμε όμως τα κράτη-μέλη να οικειώνται το κράτος δικαίου, αυτά θα πρέπει να εγγυώνται και το, ε, το, να μην υπάρχει παιδική φτώχεια. Εγώ είμαι από την Ισπανία στην Ισπανία είναι αδιανόητο να μην πηγαίνει σχολείο ένα παιδί, να μην έχει φαγητό ένα ε, παιδί, να μην έχει πρόσβαση στην υγεία ένα παιδί. Γιατί υπάρχουν ειδικέ υπηρεσίες που επιλαμβάνονται αν κάτι πάει στραβά. Κοινωνικές, λειτουργεί, ε, πρόνοια, υγεία κτλ. Για να μην συμβεί γι' αυτό αν συμβαίνει στην Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι κάπου τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ ήμουν 10 χρόνια σε μια ε, αυτοδιοίκηση περιφερειακή, και, ε, τοπική κυβέρνηση στην Ισπανία και 15 χρόνια ε, σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Όταν βλέπεις ότι ένα παιδί δεν πηγαίνει καλά, ότι ε, πάσχει από κάτι, από υποσυτισμό, από κάποια ασθένεια, επεμβαίνουν οι υπηρεσίες. Άρα όταν αυτό δεν συμβαίνει, κάτι πάει στραβά στα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να διαρθρώσουμε αυτή την παιδική, την εγγύηση μάλλον για την, ε, τα παιδιά, για να μην χαλαρώσουν τα κράτη-μέλη και αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι το οποίο ε, ε, είναι καθήκον των κρατών μελών. Συμπληρωματικέ, είπε η Επίτροπο, ότι αυτέ οι δράσει. Αλλά υπάρχουν τα διαρθρωτικά ταμεία που για αυτή τη δουλειά υπάρχουν θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι κάνουν τα κράτη-μέλη, με ποιο τρόπο εκτελούν τα προγράμματα, τι πάει στραβά για να δούμε πώς εμείς θα το συμπληρώσουμε. Γιατί καμιά φορά φοβάμαι ότι αυτή η εγγύηση για τα παιδιά θα έρθει να υποκαταστήσει κάτι που δεν κάνουν τα κράτη-μέλη. Συμπροματική να είναι η δράση μας, αλλά ε, όχι να απαλλάξουμε από τις ευθύνες τους τα κράτη-μέλη. Γιατί αυτά οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά που είναι τα πιο ευάλωτα πρόσωπα στην κοινωνία. Και η καταπολέμηση της φτώχειας ακούσαμε ε, ότι θα γίνει και από τον κοινωνικό πυλώνα. Και μια που μιλώ και για την αναπηρία. Λέμε ότι θέλουμε εκπαίδευση χωρίς ε, αποκλεισμούς. Αλλά αν δούμε το χάρτη, το σχολικό, ας πούμε, στα κράτη-μέλη, είναι ανέκδοτο αυτό ότι δεν έχει αποκλεισμούς. Σε κανένα κράτος μέλος δεν ισχύει. Γιατί η εκπαίδευση και το σχολείο είναι ένας πυλώνας που θα μας οδηγήσει σε ένα πιο δίκαιο κόσμο. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, το θέμα των παιδιών με αναπηρίες. Και ευχαριστώ πολύ τους επιτρόπους για το έργο τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντράγκος Πιτσάρου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζοντα... θα ήταν μάταιο να συνεχίσουμε να μιλάμε για τη σημασία της εγγύησης για τα παιδιά. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι σημαντική. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τη σημασία των παιδιών στην κοινωνία. Το πρόβλημα είναι αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία για να βοηθήσουμε την θεμελιώδη μεταρρύθμιση στην ε, κοινωνία μας. Μιλάμε για την ε, πράσινη συμφωνία. Γιατί να μιλήσουμε για την ε, συμφωνία για τα παιδιά και την νεολαία. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο δαπανάτε τώρα ανεπαρκώς, γιατί δεν ε, επενδύουμε στην πρόληψη, στην πρώιμη παιδική ηλικία, στην νεολαία μας και μετά έχουμε τεράστια, τεράστιους λογαριασμούς για το δημόσιο τομέα. Ένα τρεις θα μπορούσαμε να το μειώσουμε κατά πολύ με σωστά μέτρα για τα παιδιά και τους νέους. Το θέμα δεν είναι, δεν είναι αν θα προχωρήσουμε. Το θέμα είναι μπορούμε να ξεπεράσουμε τρεις διαφορές. Η μία είναι η πολιτική διαφορά, οι πολιτικές διαιρέσεις που σημαίνουν ότι ακόμα έχουμε μεγάλο διαχωρισμό μεταξύ εκείνων των ομάδων που πιστεύουν σε δικαιώματα και στη νομική υποχρέωση των κρατών να χειριστούν τα δικαιώματα, πολύ σημαντικό, και άλλη ομάδα που ε, θεωρεί τις επενδύσεις το κρίσιμο ζήτημα. Τώρα όμως έχουμε αποδείξεις ότι ε, οι επενδύσεις ε, δεν μπορεί να έχουν και κοινωνική οικονομική απόδοση όπως η οικονομική. Θα πρέπει να τα συνδυάσουμε. Έτσι θα ξεπεράσουμε αυτή τη ε, διαφορά. Επίσης, διαφορά μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού. Υπάρχει η τάση να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να είναι υπόλογο μόνο στο τομέα. Όχι. Υποκρισία. Θα πρέπει να έχουμε μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Κρίσιμο θέμα αυτό. Τέλος, η διαφορά σε σχέση με τη διακυβέρνηση. Μπορεί να τα γνωρίζουμε αυτά σε, τοπικό, σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά πρέπει να δούμε και την τοπική αυτοδιοίκηση και να ενταχθεί. Δεν μπορεί το πρόβλημα να λυθεί αν δεν συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλίσια Χομσκιμέλ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, Ακούγοντας τις διάφορες παρεμβάσεις, η ε, κυρία Χόμς Χινέλ, ε, συμφωνούμε ότι η παιδική φτώχεια είναι μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Το ένα στα τέσσερα παιδιά κινδυνεύει να πέσει στη φτώχεια και ένα στα δέκα είναι ήδη στον κοινωνικό αποκλεισμό. Ε, θα πρέπει πολύ νωρίς ε, να φροντίσουμε να μην χάνονται ευκαιρίες των παιδιών. Ε, είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ ότι το Δεκέμβριο του 2018 συμφωνήσαμε το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ θα πρέπει να δώσει 5,9 ε, δις για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Βέβαια, και στο μελλοντικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντανακλάται αυτό. Την περασμένη Παρασκευή είδαμε την πρόταση για τη διαπραγμάτευση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με κάποιες περικοπές σε πολύ σημαντικούς τομείς για την κοινωνική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι είναι κάπως ανησυχητικό αυτό. Και δεν προμηνεί ε, πολλά θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη αυτό το πρόβλημα, αλλά χρειάζεται και ευρωπαϊκή βοήθεια, οικονομική βοήθεια, γιατί παρατηρείται παντού όπως είπαμε. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να κάνουμε περικοπές στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φαπιόλα Κερδός από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω σε αυτό το εγχείρημα το οποίο αφορά ανθρώπους και μάλιστα παιδιά και όχι αριθμητικά στοιχεία. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον πράγματι. Άκουσα τον αντιπρόεδρο που μίλησε, την αντιπρόεδρο που μίλησε για την δημοκρατία και πραγματικά υπάρχει εδώ μια ευτυχή σύνδεση ότι στην ίδια Επιτροπή ε, βρίσκονται δύο εξίσου σημαντικά θέματα που μας επιτρέπουν να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια αλλά και να βελτιώσουμε τα δημογραφικά στοιχεία και την ένταξη στην Ευρώπη. Τώρα, η εγγύηση για το παιδί. Ε, αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο για την επίτευξη και των δύο στόχων. Και αν με τους δύο στόχους μεταξύ μας, ερωτώ, υπάρχουν μέτρα που διαφοροποιούν τα θέματα στις επιμέρους χώρες μέλη, γιατί στις χώρες μέλη υπάρχει ακόμα μεγάλη διαφορά μεταξύ αγοριών κοριτσιών. Πώς μπορούν να ρυθμιστούν αυτά. Υπάρχουν και μέτρα διαφοροποίησης όταν πρόκειται για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ε, ταυτότητα του φύλου. Υπάρχουν επίσης μέτρα για την καταπολέμηση της βίας που ασκείται σε πολλές χώρες κατά των παιδιών αυτών. Ευχαριστώ. από την Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροποι, κυρίες και κύριοι. Μας ενδιαφέρει πολύ η σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία για την εγγύηση για τα παιδιά. Επίσης, άκουσα με χαρά για τη συνάντηση με τον κύριο Σμιτ στην Πολωνική Βουλή και τον ευχαριστώ πολύ για τη συνάντηση. Η στήριξη των οικογενειών και η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας είναι από τις μεγάλες προτεραιότητες της πολωνικής κυβέρνησης. Από τον Απρίλιο του 2016 αρχίσαμε ε, πρόγραμμα στήριξης οικογενειών με παιδιά. Αυτό είναι κομμάτι ε, ενό προγράμματο που λέγεται Οικογένεια 500 ΣΥΝ, η μεγαλύτερη μεταφορά χρημάτων σε πολωνικές οικογένειες από το 1989. Το πρόγραμμα Οικογένεια 500 ΣΥΝ στοχεύει στη βελτίωση της δημογραφικής κατάστασης, μειώνει τη φτώχεια μεταξύ των νέων και είναι επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο ε, θεσπίσαμε στην Πολωνία είναι ένα πρόγραμμα για ανθρώπους μεταξύ 7 και 20 ετών που εκπαιδεύονται. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία μέχρι, ηλικίας μέχρι 25 ετών, 24 ετών και εδώ φροντίζουμε να τους δώσουμε καλή, μια καλή αρχή στη ζωή. Επίσης, ε, στοχεύουμε στην αύξηση της πρόσβασης ε, στη φροντίδα, σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας για παιδιά μέχρι 6 ετών. Επίσης, έχουμε και άλλο πρόγραμμα στήριξη οικογενειών και παιδιών. Είναι μια κάρτα μεγάλη οικογένεια για να στηρίξει πολλές οικογένειε με παιδιά και τους επιτρέπει να ωφεληθούν από κάποιες εκπτώσεις σε καταστήματα και αλλού. Η κάρτα της μεγάλης οικογένειας είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των οικογενειών και πάνω από 6.500 ε, οικογένειες συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό με τις εκπτώσεις και την υποστήριξη. Κάτι άλλο ε, τέλος κυρίες και κύριοι. Αυτές ε, είναι πρωτοβουλίες σημαντικές που πρέπει να τις ε, δούμε και να κοιτάξουμε και το θέμα του, της βίας και των ε, προβλημάτων με το διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, συμμετασχόντες στη συζήτηση. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη και θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν για τη δική του συνεισφορά. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα και χαίρομαι που σε όλες μας τις συζητήσεις συμφωνήσαμε στην προώθηση αυτού του θέματος. Όλοι συμφωνούμε πώς θα γίνει αυτό. Είναι κάτι πολύ λογικό. Όλοι οι άνθρωποι, όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία εμείς πρέπει να φροντίσουμε να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Πολλά θα ακούσουμε ακόμα για τις νέες πρωτοβουλίες. Έχετε την πλήρη υποστήριξή μου και πράγματι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η Κομισιόν και όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χειριστούν το θέμα όσο γίνεται πιο σοβαρά και εμείς από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και ε, στην ε, υλοποίηση των ονείρων τους, ανεξάρτητα από το που ζουν και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συμβεί αυτό. Είμαι πεπισμένος ότι το πρόβλημα θα λυθεί και μάλιστα στο εγγύς μέλλον. Τώρα θέλω να δώσω το λόγο ε, στην ε, κυρία Νίκολ Σόνοβα. Περνάμε τώρα στη δεύτερη συνεδρία για, τους, ε, για τον δίκαιο κατώτατο μισθό. Από όλη τη συζήτηση όμως που έγινε μέχρι τώρα, μοιάζει ότι αυτό συνδέεται με την εγγύηση για τα παιδιά. Είπε ο Επίτροπος ο κύριος Σμίτ ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για να ενισχυθούν οι γονείς βοηθούν και τα παιδιά. Θα ήθελα λοιπόν αρχικά να δώσω το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Σμιτ, για μια σύντομη παρουσίαση του θέματος των, ε, του δίκαιου κατώτατου μισθού. Adequate wages are είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, το δίκαιο κατώτατο του μισθού, για να υπάρχουν σωστές συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς διαβούς διαβίωσης ε, για όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εργαζομένους. Αυτό τονίζεται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, είναι αρχή υπαριθμών 6. Ο κατώτατος μισθός είτε ε, ορίζεται από τον νόμο είτε από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι εκ των όνου κάνευ για να προστατεύει τους μισθούς. Αυτό το κάνει κατώτατη μισθή για να ε, αποτρέψουμε ε, τα φαινόμενα εργαζομένων φτωχών και ανισοτήτων. Θα πρέπει να πιάνει τόπο η δουλειά, να αμείβεται σωστά και να ενισχύεται η συμμετοχή και των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, οι επιδόσεις διαφέρουν πάρα πολύ από χώρα σε χώρα και μάλιστα και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Οι ανισότητε στους μισθούς έχουν αυξηθεί. Η ψαλίδα αυτή έχει ανοίξει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση παντού, όπου πολλοί χαμηλά αμοιβόμενοι έχουν δει να μειώνεται η αγοραστική τους δύναμη ε, συγκριτικά με άλλες ομάδες κοινωνικές. Ε, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη νέα υπόσχεση ε, των ευρωπαϊκών ε, προγραμμάτων για την πρόοδο και την ευημερία. Γι' αυτό η κυρία Φόντερ Λάιεν πρότεινε και παραθέτω να προταθεί ένα νομικό μέσο ε, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα δίκαιο κατώτατο μισθό. Υπό την έννοια αυτή στις 14 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκρινε ένα έγγραφο το οποίο λανσάρει τον πρώτο γύρο, τη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων για την ανάγκη και την ενδεχόμενη κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η ευρωπαϊκή δράση για κατώτατους μισθούς. Μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δίκαιους κατώτατους μισθούς θα συνεισέφερε πρώτον στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης χαμηλά αμοιβωμένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να τονωθεί η ζήτηση ε, διατηρώντας ε, την ανταγωνιστικότητα αλλά και την εργασία. Δεύτερο στόχος, σύγκληση προς τα πάνω σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας σε όλα τα κράτη-μέλη και στη δημιουργία ε, ισότιμων κανόνων παιχνιδιού για τις επιχειρήσεις σε μια ενιαία αγορά. Και στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα πολιτική ορμή υποστηρίζοντας ε, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες στα κράτη-μέλη. Είναι σαφές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δεν πρόκειται, δεν πρόκειται να επιβάλλει ένα νομιόμορφο κατώτατο μισθό σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε πρέπει να γίνει. Ε, αυτό θα είχε επιπτώσει στην απασχόληση και στην οικονομική ευρωστία. Μια τέτοια πρωτοβουλία επίσης δεν πρόκειται να επιβάλλει επίσημο θεσμικό κατώτατο μισθό σε χώρες που έχουν μεγάλη κάλυψη από τις συλλογικέ συμβάσεις και διαπραγματεύσεις. Τα συστήματα αυτά δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τις διατάξεις αυτές αρνητικά. Θα υπάρχει εγγύηση και προστασία τους. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε χώρες όπου αυτές είναι αδύναμες. Άρα ε, έχει στόχο να προάγει τον κοινωνικό διάλογο και ε, τις ε, θεσμική διάσταση της κοινωνικής συμμετοχής. Οι κατώτατοι μισθοί θα εξακολουθούν να ορίζονται είτε με νόμο είτε με τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις με πλήρη σεβασμό της εθνικής παράδοσης και της αυτονομίας δράσης των κοινωνικών εταίρων. Ε, λανσάραμε την πρώτη φάση διαφουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Στη συνέχεια, η φάση αυτή ολοκληρώνεται τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου περίπου, και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τις απόψεις που θα έχουν καταθέσει οι κοινωνικοί εταίροι και θα αφήσει τους κοινωνικούς εταίρους να αποφασίσουν ε, αν θα προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λανσάρει τη δεύτερη φάση διαβουλεύσεων έτσι ώστε να ε, συζητήσουν το ενδεχόμενο περιεχόμενο ε, της πρωτοβουλίας για κατώτατους μισθούς, δίκαιους κατώτατους μισθούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Στεριανή Μπιζίου. Ελπίζω να πρόφερα καλά το όνομά σας, λέει η πρόεδρος. Είναι λίγο δύσκολο για μένα. Είναι μέλος της ε, Μόνιμης Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Έχετε το λόγο. Πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντε Λάιεν, για την τόσο κέρια και ευιστοποιημένη πρωτοβουλία που ανέλαβε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατοχυρώσει δίκαιε και αξιοπρεπείς συνθήκε διαβίωση για όλου του εργαζόμενου. Απαραίτητο εργαλείο και πρώτο βήμα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η θέσπιση του κατώτατου μισθού. Και ω γυναίκα προσδοκώ ότι θα συντελέσει στην μείωση, αν όχι στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματο, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμη ανάμεσα στα δύο φύλλα. Στην Ελλάδα, ο κατώτατος μισθός, όπως και το ημερομίσθιο, ρυθμίζονται με νόμο ήδη από το έτος 2012. Πριν το 2012 και ήδη από το 1998, ο κατώτατος μισθός ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Με νόμο του 2013 εισήχθη το ισχύον σύστημα ορισμού του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου μερομισθίου που προβλέπει ευρεία διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και τη κυβέρνηση με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών και συναφών φορέων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα οικονομίας, της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής και εργασιακών σχέσεων. Σύμφωνα με την τρέχουσα ελληνική νομοθεσία, το ύψος του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και των μισθών. Η συγκεκριμένη διαδικασία ξεκίνησε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2019 με την έκδοση υπουργικής απόφασης βάσει της οποίας καθορίστηκε ο νόμιμος κατώτατος μισθός στα 650 ευρώ. Για να γίνει κατανοητή η αγοραστική δύναμη του ποσού αυτού, θα αναφέρω ότι ένα φθηνό γεύμα στην Ελλάδα κοστίζει 10 ευρώ, όσο δηλαδή και στη Βουλγαρία, ενώ στο Λουξεμβούργο κοστίζει σχεδόν 17 ευρώ. Το ενίκιο ενός μικρού διαμερίσματος ξεπερνά τα 300 ευρώ, ενώ στη Βουλγαρία ανέρχεται στα 270 ευρώ και στο Λουξεμβούργο το ίδιο διαμέρισμα φτάνει τα 1.500 ευρώ. Και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα τις δύο αυτές χώρες, διότι αντιστοιχούν στον χαμηλότερο και υψηλότερο κατώτατο μισθό στην Ευρώπη αντιστοίχω. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1998 έως το 2011 ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αυξανόταν συνεχώς, με την τελευταία αύξηση να γίνεται τον Ιούλιο του 2011. Τον Μάρτιο του 2012, ο κατώτατος μισθός μειώθηκε κατά 22% για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών και κατά 32% για τους εργαζόμενους από 18 έως 25 ετών. Η μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα της κρίσης χρέους και των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Ο κατώτατος μισθός και η αύξησή του εντός του 2020 είναι στην ελληνική επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα συνδέεται και με διάφορα επιδόματα, τα οποία θα αυξηθούν και αυτά εντό του έτους ως συνέπεια αύξησης του κατώτατου μισθού. Από την πιθανή αύξηση θα επηρεαστούν περίπου 700.000 μισθωτοί, που είτε εισπράττουν τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ με πλήρη απασχόληση, είτε εργάζονται με καθεστώ μερική απασχόληση και λαμβάνουν ω μισθό κάτω από 500 ευρώ και γενικότερα όσοι εξαρτώνται ευθέω από το ύψο του κατώτατου μισθού. Σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργό μα επεσήμανε πω η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ τη αύξηση του κατώτατου μισθού, που πρέπει όμω να συνδέεται με το ρυθμό τη οικονομική μεγέθυνση και την παραγωγικότητα τη οικονομία μα. Το θέμα του κατώτατου μισθού απασχολεί διαχρονικά την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την οικονομική και εργασιακή ανάπτυξη, την καταπολέμηση των μισθολογικών ανισοτήτων και της εργασιακής φτώχειας. Η Ελλάδα στέκεται αναμφισβήτητα υπέρ του ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού. Η ελληνική θέση είναι να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό, ο οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε εθνικό νομοθέτη να ορίζει τον κατώτατο μισθό βάσει των ιδιωτεροτήτων του εσωτερικού εθνικού δικαίου, των προβλέψεων και των στοιχείων τη εθνική οικονομία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προάγει και ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο και τι δημοκρατικέ διαδικασίε. Οι οικονομικές πολιτικές της Ελλάδας έχουν έντονο κοινωνικό περιεχόμενο με στόχο τη θωράκιση του εισοδήματος των εργαζομένων και την προστασία της εργασίας στο πλαίσιο σύγχρονων και αποτελεσματικών πολιτικών. Η στάση της Ελλάδας είναι τόσο φιλοεπενδυτική όσο και φιλεργατική, καθώς το ένα προάγει το άλλο οποιαδήποτε δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των κατώτατων μισθών, σεβόμενη τι εθνικέ παραδόσει, την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και την ελευθερία των διαπραγματεύσεων, είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Εν κατακλείδη, η ουσία των δράσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται στου δυσνόητου όρου και τι συντομογραφίε, αλλά στον αντίκτυπο που έχουν αυτέ στην καθημερινότητα του εργαζόμενου. Στόχο όλων μα είναι οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν εξασφαλισμένο ένα δίκαιο μισθό, ο οποίος θα είναι επαρκής για έναν αξιοπρεπή τρόπο διαβίωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει τώρα η συζήτηση μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Long list of speakers and... Είναι μακρύς ο κατάλογος των ομιλητών, αλλά ο χρόνος περνάει. Ξέρετε ότι πρέπει να τελειώσουμε στις 7 ακριβώς θα σας παρακαλούσα πώς να το πω, να φροντίσετε ε, το χρόνο σας ε, να τον τηρείτε. 1,5 λεπτό έκαστος. Ζητώ συγγνώμη, αλλά τι να κάνω. Η κυρία Άννα Γιωχάνσον από τη Σουηδία, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ε, ότι καλωσορίζω τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει μια βιώσιμη Ευρώπη με καλές συνθήκες εργασίας για όλους. Ε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό όμως τι σημαίνει. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι εθνικές αρμοδιότητες. Διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ο κατώτατος μισθός είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Όπως σας είπαμε, ενησυχούμε βαθύτατα από την όλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει ε, ε, ε, δεν θέλουμε να μας αναγκάζεται να προχωρήσουμε σε νομιθωτικές αλλαγές. Είναι πολύ σημαντική η αυτορύθμιση και η δυνατότητα κάθε κράτους μέλους να προχωρεί σύμφωνα με τις παραδόσεις. Εδώ πρόκειται για ολόκληρη την αγορά εργασίας, τους μισθούς. Είναι πολύ διαφορετικά τα μοντέλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι εξασφαλίζει κάθε χώρα τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητά της. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Εμείς είμαστε κατά της οδηγίας ε, και η ε, οικονομία στη χώρα μας αλλά και το συνδικαλιστικό κίνημα και τα διάφορα πολιτικά κόμματα στην Σουηδική Βουλή είναι αντίθετα με τις κατευθυντήριες γραμμές αυτές της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Έχουμε προβλήματα και με τις συστάσεις. Δεν θέλουμε να μας περιορίσετε τις δυνατότητες που έχουμε να παίρνουμε ε, μέτρα με βάση τη σουηδική αγορά εργασίας. Ε, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να κοιτάξουμε τα λογικά μέτρα που χρειάζονται σε όλη την Ευρώπη. Η κυρία Σφετλάνα Αγγέλοβα από τη Βουλγαρία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ε, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ε, ε, είναι ο κατώτατος μισθός, αυτό που μας απασχολεί σήμερα το θέμα, πολύ σημαντικό για την Βουλγαρία. Όχι μόνο γιατί έχουμε σοβαρές δημογραφικές προκλήσεις, αλλά και γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε υψηλό βιωτικό επίπεδο για όλους τους κατοίκους της χώρας. Για το λόγο αυτό στην ε, Βουλγαρία έχουμε ξεκινήσει μια ευρύτατη διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, το Νοέμβριο θα δώσουμε τη συνεισφορά της Βουλγαρίας για το πρόγραμμα δράσης για το πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Βουλγαρία είναι από εκείνα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ε, Υπάρχει ρύθμιση για τον κατώτατο μισθό βασιζόμενη ε, στις ανάγκες και στις ε, πραγματικότητες της οικονομίας αλλά και στις δυνατότητες των εργοδοτών. Για μας είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι αποτελεί αυτό μια καλή βάση για οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε εθνικό επίπεδο και έχουν αυξηθεί και οι συνθήκες εργασίας και το βιωτικό επίπεδο. Ένας δίκαιος κατώτατος μισθός είναι ένα πολύ καλό θέμα για την ευρωπαϊκή αυτή διαβούλευση. Θα αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο και θα υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα, ο κύριος Ντάνιελσον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σένα, Νίκολας, για την εισαγωγή σου. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα του, ε, των ευρωπαϊκών κατώτατων μισθών. Ακούσαμε και από τη συνάδελφο από τη Βουλή της Σουηδίας ε, ότι υπάρχουν δισταγμοί ε, για την οδηγία. Θα προτιμούσαμε συστάσεις να απευθύνεται και όχι οδηγία. Αλλά θέλω να πάω αλλού λίγο τη συζήτηση. Εχθές ε, στην Επιτροπή μας συζητήσαμε με το, τη Eurofound τους, ε, το θέμα των εργαζομένων φτωχών. Αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο να είναι εργαζόμενοι φτωχοί είναι αυτοί που εργάζονται με μερικό ωράριο, αυτοαπασχολούμενοι, ε, ε χωρίς να το επιθυμούν οι ίδιοι, έχουν διαφορετικά είδη ε, συμβάσεων προσωρινής εργασίας. Το ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, αλλά τι μπορούμε εμείς να κάνουμε μαζί με την πρωτοβουλία για τους κατώτατους μισθούς, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να επιλέγει, ε, έστω και αν είναι προσωρινή εργασία, να είναι πλήρους απασχόλησης και όχι αυτές τις άτυπες μορφές εργασίας, γιατί συνδέονται πάρα πολύ με την έννοια του εργαζόμενου φτωχού. Ευχαριστώ. κυρία Μάρα Καλίστα από την ε, Ρουμανία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Ρουμανία κοιτάζει με ανυπομονησία, την, περιμένει με ανυπομονησία την, απόφαση για το θέμα αυτό. Και χαιρόμαστε που σέβεστε τις εθνικές αποφάσεις δεδομένου των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Η Ρουμανία είναι μια από τις χώρες που έχει έναν νομικά κατοχυρωμένο κατώτατο μισθό, αλλά διαρωτώ με τι συμβαίνει όταν δεν συνεννοούνται οι κοινωνικοί εταίροι. Εδώ αναφέρομαι στα συνδικάτα και τους εργοδότες. Μερικές φορές συμβαίνει και αυτό. Τι συμβαίνει όταν δεν μπορούν να διαπραγματευτούν με ώστε να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Μήπως θα πρέπει να σκεφτόμαστε κάποιο νομοσχέδιο που θα αφορά τους κατώτη, τον κατώτατο μισθό και αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του μόνο τα οικονομικά στοιχεία όπως την παραγωγικότητα και άλλα γιατί η αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να τα αποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα κάθε χώρας. Κάθε χώρας. Το λέω αυτό και υπογραμμίζω ότι στη Ρουμανία, παραδείγματος χάρη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξασφαλίζουν το 58% του ΕΠ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικές οι μετρήσεις που γίνεται και η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα δοθεί για να μην καταστραφεί ο ιδιωτικός τομέας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγγες Βεσέλης από τη Μάλτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά και προτείνει αυτό το πλαίσιο του κατώτατου μισθού για όλα τα κράτη-μέλη. Η Μάλτα ήδη έχει νόμιμο κατώτατο μισθό που καλύπτει όλους τους εργαζομένους. Το 2017 έγινε αναθεώρηση του κατώτατου μισθού. Συμφωνήθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό για διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Μετά από αυτό το διάστημα πρέπει να τους δοθεί αύξηση. Αύξηση στο βασικό τους μισθό. Ακόμα λοιπόν και αν υπάρχει, παρότι υπάρχει νόμος για τον κατώτατο μισθό, αυτός δεν μπορεί να καταβάλλεται σε έναν εργαζόμενο για μεγαλύτερο διάστημα ε, αυτό έχει γίνει αυτό έχει αυξη... ο κατώτατος έχει αυξηθεί για πέντε συνεχόμενα έτη χωρίς παράλληλη αύξηση των φόρων. Τώρα, όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, γνωρίζουμε και υπάρχουν προγράμματα ε, που βοηθούν τα άτομα αυτά να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και με τα προγράμματα αυτά πολλοί έχουν αποκτήσει τέτοια πρόσβαση. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι, λίγοι, που ακόμα και με τη βοήθεια των προγραμμάτων δεν έχουν αρκετές δυνατότητες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Χρειάζονται όμως αξιοπρέπεια. Προς χάρη αυτών λοιπόν θα, θα, θα δοθεί ένας κατώτατος μισθός σε αυτούς για να ζουν με αξιοπρέπεια. Τα άτομα λοιπόν αυτά με σοβαρές αναπηρίες θα, θα έχουν ένα επίδομα που θα είναι αντίστοιχο του κατώτατου μισθού. Ε, έχετε, ε, έχετε, έχει περάσει ο χρόνος η κυρία Μπίσοφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ παιδική φτώχεια και ελάχιστη μισθή. Αυτά τα δύο θέματα είναι συνειφασμένα. Αν δεν υπάρχουν ε, ελάχιστη μισή θα υπάρχει παιδική φτώχεια. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να καταπιαστούμε με το θέμα και είμαι ευγνώμων που το κάνει η Κομισιόν και έχει το απαραίτητο θάρρος. Και είδαμε, τόπικη συνάδελφος, ότι είχαμε τη στρατηγική 2020 που θέλαμε οπωσδήποτε να μειώσουμε τη φτώχεια. Δεν λειτουργήσε το σύστημα, αυξήθηκε η φτώχεια. Τώρα προχωρούμε με σοβαρότητα. Αναλαμβάνουμε δέσμευση. Αυτό είναι σημαντικό βήμα. Αλλά ακούμε επίσης ότι υπάρχουν διαφορετικές στάσεις γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν πολλούς φτωχού, που εργάζονται και φτωχοί και υπάρχουν και άλλοι που έχουν ε, διαφορετική ε, πολιτική και μπορούν να διασφαλίσουν το πρόβλημα ε, χωρίς εργασία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την πολιτική ε, ε, των τιμών, εκεί που είναι ισχυρή αλλά και εκεί που είναι αδύναμη βέβαια, γιατί η ελάχιστη μισθή είναι η πιο χαμηλή προσέγγιση. Αλλά το να υπάρχουν καλοί μισθοί σε, στην Ευρώπη, σε μια ανθυρή ήπειρο, Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε. Στην, ε, ε, έχουμε και, ε, ε, στοιχεία και για την Ελλάδα που είναι αρνητικά. Πρέπει να προσεγγίσουμε ότι όλοι πρέπει να δουλεύουν και να ε, ωφελούνται από την εργασία του. Ευχαριστώ κύριος Μπάρτσα από την Ουγγαρία. Το Ουγγρικό Κοινοβούλιο παρακολουθεί πολύ στενά τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα δίκαιο κατώτατο μισθό. Χαιρόμαστε που ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σεβαστεί τις συλλογικές συμβάσεις, τις παραδόσεις κάθε χώρας και ε, ε, τα ε, όσα παραδοσιακά συμβαίνουν. Ελπίζω οι ε, βουλευτές από τη χώρα μου να συμμετέχουν στη συζήτηση. Διπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια ο τους μισθός για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει μειωθεί και η ψαλίδα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ανησυχούμε ήδη σε ό,τι αφορά την νομική βάση, αλλά και τις αρμοδιότητες ε, των κοινωνικών εταίρων. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της ε, την ε, ε, διαβούλευση, το αποτέλεσμά τη και να κάνει σε βάθο μελέτη επιπτώσεων. Όλοι γνωρίζουμε ότι στο παρόν οικονομικό πλαίσιο Ανεβαίνουν παντού οι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και χωρίς επέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως στις χώρες της ε, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως διαβάζουμε στη σχετική έκθεση για την εργασία. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι εθνική αρμοδιότητα και διαφέρουν πολύ οι πραγματικότητες. Η κυρία Σντανόκα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Yes. Η πολιτική μας ομάδα, η ομάδα ΓΚΟΕ, εργάστηκε πολύ και έδωσε μάχες για να υπάρχει μια ενιαία θέση στον κατώτατο μισθό και το ελάχιστο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω το ψήφισμά μας από τον Απρίλιο 2019 όπου μιλήσαμε για ελάχιστο εισόδημα. Κύριε Σμιτ, Σμιτ ελπίζουμε ειλικρινά η Κομισιόν όταν καταπιαστεί το θέμα του ελάχιστου μισθού δεν θα ξεχάσει και το ελάχιστο εισόδημα σε επίπεδο ένωσης γιατί ιδιαίτερα η παιδική φτώχεια και η καταπολέμησή της έχει περισσότερη σχέση με το ελάχιστο εισόδημα και όχι με τον ελάχιστο μισθό. Όταν μιλάμε για τον ελάχιστο μισθό, ανησυχούμε διότι προτείνεται να μην πάρουμε τον μέσο αλλά τον διάμεσο μισθό. Και αυτό είναι διαφορετικό, δηλαδή συνεπάγεται μεγάλες διαφορές μισθών. Αλλά θα το συζητήσουμε και αργότερα αυτό, αργότερα. Ε, Ο κύριος Λάσλο Βάριο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Κύριε Πίτροπε, Υποστηρίζουμε τις ε, πρωτοβουλίες υπέρ μια ισχυρής Ευρώπης. Συμφωνώ με όλα αυτά που λέτε, ότι στην Ευρώπη χρειαζόμαστε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να την αδράξουν αυτή την ευκαιρία. Σε ό,τι αφορά τις διάφορες κοινωνικές πρωτοβουλίες, η βάση τους μπορεί να είναι μια ισχυρή οικονομία. Από την άλλη, δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε ισχυρή οικονομία παρά μόνο εάν είναι ε, σωστές οι κοινωνικές προϋποθέσεις. Οι δεξιότητες, η εκπαίδευση, η κατάρτιση των εργαζομένων καθορίζουν το ίδιο το καθεστώς της οικονομίας. Στην Ουγγαρία έχουμε 4,4 εκατομμύρια πολίτες και το 3,1 εκατομμύρια αμείβονται με μισθό κατώτερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε λοιπόν υπέρ του κατώτερου μισθού. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν αντίστοιχε εμπειρίες και θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την πρωτοβουλία, ιδιαίτερα στο διάλογο και τη διαβούλευση ε, με τους κοινωνικούς εταίρους και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ξέρετε ότι σχολάνε οι διερμηνήσεις 7 ακριβώς. Έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές. Μειώνω το χρόνο από ένα και, ε, λεπτό και μισό σε ένα και είκοσι δεύτερα. Είναι πολύ σκληρό για μένα, αλλά τι να κάνω. Ε, επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Ντεμιρέλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης στο άρθρο 4 προβλέπει το δικαίωμα για δίκαιη αμοιβή εργασίας και σε αυτό το χάρτη ρυθμίζεται σαφώς ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να παίρνουν αξιοπρεπή μισθό για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Βέβαια, τι σημαίνει κατάλληλος μισθός ή δίκαιος μισθός. Γίνονται συζητήσεις, αλλά το ελάχιστο που αποκλείει τα δύο κριτήρια είναι ότι οι ε, άνθρωποι που εργάζονται έχουν μισθούς φτώχειας και ξέρουμε και έχουμε ορισμό τι είναι η φτώχεια. Το 60% του μέσου εισοδήματος ορίζεται αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άνθρωποι που είναι κάτω από το 60% ε, απειλούνται από τη φτώχεια. Ε, αν ε, δούμε και θέλουμε να τηρήσουμε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη, αυτό ορίζεται ξεκάθαρο τι είναι ο ελάχιστος μισθός, που είναι το 60% του διάμεσου μισθού. Ε, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη έχουν ελάχιστο μισθό. Εγώ είμαι από την Γερμανία και εμείς έχουμε ελάχιστο μισθό, αλλά είναι τόσο χαμηλός που οι άνθρωποι που παίρνουν αυτό το μισθό αργότερα ε, έχουν ε, ε, φτώχεια κατά την τρίτη ηλικία τους μετά τη συνταξιοδότηση. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε σαφές, σαφείς δεσμεύσεις και να ε, έχουμε σαφή ορισμό σχετικά με το τι είναι φτώχεια και τι προστατεύει από αυτήν. Και τέλος, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να κάνει πολιτική μισθών. Δεν πρόκειται περί αυτών. Πρόκειται για την προσαρμογή των συνθήκων διαβίωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Τουραφεράντες, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ θα μιλήσω λίγο ως βουλευτής και λίγο ως Ισπανίδα. Γιατί η Ισπανική κυβέρνηση δεν μπόρεσε να στείλει Ισπανούς βουλευτές γιατί ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί σε σώμα οι κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Να σας πω λίγο πώς έχει η κατάσταση στην Ισπανία. Τα ξέρετε όλοι. Οι σοσιαλιστές κυβερνούν σε συνασπισμό με την αριστερά και έχουν δεσμευτεί για το κατώτατο μισθό. Ε, υπάρχει κατώτατος μισθός, ε, θα αυξηθεί έτσι ώστε να φτάσει στο 60% που έλεγε η ε, προλαλήσασα και το, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας και ο Κοινωνικός Χάρτης και με τη συμφωνία των εργοδοτών. Αυτό που συμβαίνει τι είναι τώρα. Είναι γεγονός ότι ένας κατώτατος μισθός που ορίζεται δια νόμου από την κυβέρνηση ε, μπορεί να αλλάξει όταν αλλάξει η κυβέρνηση και έρθει άλλο κόμμα. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κοινωνική και κοινοτική ε, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Σίγουρα δεν πρόκειται να εκριζωθεί η φτώχεια αν έχουμε κατώτατο μισθό, αλλά είναι ε, εκ των όνων κάνευ για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και από την Ισπανία πρέπει να σας πω ότι η σοσιαλιστική ομάδα ε, υποστηρίζουμε μία πρωτοβουλία που ενισχύει φυσικά ε, τι συλλογικέ διαπραγματεύσεις και τι συλλογικέ συμβάσεις και τη θέση των εργαζομένων, αλλά και αξιοπρεπείς μισούς σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Ντένις Ράτκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε. Έχετε αναλάβει δύσκολο καθήκον πραγματικά γιατί το θέμα ελάχιστος μισθό. Ε, δεν είναι μόνο ένα που ενδιαφέρει πολύ και προσελκύει πολλές συζητήσεις, αλλά ε, συνεπάγεται και πολλά προβλήματα που τα ε, παρουσίασε η πρόεδρος της Επιτροπής. Στις πρώτες 100 μέρες πρέπει να υπάρχουν προτάσεις. Ε, εσείς πάντως θα έχετε και την αξίζετε κάθε στήριξη και συνάδελφοι από τις βόρειες χώρες ε, ζήτησαν το λόγο. Αντιλαμβάνομαι τις επιφυλάξεις τους γιατί στις βόρειες χώρες αλλά και στην Αυστρία υπάρχουν λειτουργικά καλά συστήματα και ανησυχούν εκεί τι ε, επιπτώσεις θα υπάρξουν στο δικό τους το, στα δικά τους συστήματα. Σε όλη αυτή τη συζήτηση δεν πρέπει να δούμε όμως τι ποιο σύστημα λειτουργεί, αλλά να δούμε και τι, που δεν λειτουργεί το σύστημα και όπου, υπάρχει παράδοση κοινωνικών εταίρων και ε, όπου δεν υπάρχει καθόλου. Και γι' αυτό προσκαλώ τα κράτη-μέλη που έχουν λειτουργικό σύστημα να βοηθήσουν ούτω ώστε να έχουμε λειτουργικά συστήματα και εκεί που δεν υπάρχουν τώρα. Η κυρία Τζάντερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η τελευταία μας ομιλήτρια. Με Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Ήθελα φυσικά και εγώ να καλωσορίσω και να χαιρετήσω όλες τις πρωτοβουλίε που στρέφονται προς περισσότερη κοινωνική Ευρώπη, οι οποίοι είναι απολύτως απαραίτητοι για να προστατεύονται οι πιο ευάλωτοι, τα παιδιά, τα οποία συζητούσαμε προηγουμένως, αλλά να έχουμε και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη ε, μεταξύ των εργαζομένων των διαφόρων κρατών μελών. Και επίσης, μια φορά, για να έχουμε και περισσότερο θεμητό ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά. Επιλέξατε να ε, αφιερωθείτε, γιατί το επιλέξατε, σε αυτό το κατώτατο μισθό ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα θα είναι δύσκολο το έργο σας. Ακούσαμε σήμερα τις αντιδράσεις, γνωρίζουμε τις θέσεις των διαφόρων εδώ στο Κοινοβούλιο. Ποια είναι η δυσκολία? Το να σεβόμαστε ταυτόχρονα την αρχή της επικουρικότητας και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και να έχουμε ταυτόχρονα μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Απλή λοιπόν η ερώτησή μου. Έχετε σκεφτεί τίποτα άλλο, κανένα άλλο εργαλείο για τη μεγαλύτερη κοινωνική σύγκληση πέραν του κατώτατου μισθού που είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ πολύ. Για να κλείσουμε, όλοι βλέπουμε τη σχέση μεταξύ δίκαιου κατώτατου μισθού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη εγγύηση για τα παιδιά. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται εγγύηση για τα παιδιά, αλλά δεν συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός. Οπότε αυτό είναι μια πρόκληση, μεγάλη πρόκληση για τον κύριο Σμιτ και όλη την ε, Επιτροπή. Τώρα, δύο ανακοινώσεις πρέπει να κάνω. Ελπίζω ότι οι διερμηνείς θα μεταφράσουν. Πρώτον, θα σας συνοδέψουν από την αίθουσα συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό Σπίτι Ιστορίας όλοι συνάδελφοι και δεύτερον μην αφήσετε τίποτε προσωπικό σας στην αίθουσα αυτή γιατί όταν φύγετε από το κτίριο δεν μπορείτε να ξαναμπείτε. Πάρτε λοιπόν όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα μαζί σας. Ευχαριστώ.